είμαστε ενημερίσει σε διάταξη και πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε καθυστερήσει περιπτώσει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και του κράτους δικαίου βάσει το άρθρο 135 του κανονισμού. Θα αρχίσουμε λοιπόν με την κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα δώσω το λόγο στους συντάκτες. Ο κύριος Τάνοκ πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, το σημερινό ψήφισμα. Ε, ιδιαίτερα επικεντρώνεται στα προβλήματα των ατόμων με αφισμό, ιδιαίτερα στο Μαλάουι, αλλά το πρόβλημα είναι γενικότερο στην Αφρική. 98% των ε, ατόμων με αλφισμό πεθαίνουν πριν να φτάσουν τα 40 χρόνια ζωή στην Αφρική και λόγω τρομερών καρκίνων του δέρματος αλλά και λόγω των ε, βίων επιθέσεων που υφίστανται άτομα με αλφισμό. Ε, μόνο στο Μαλάουι 65 βία επεισόδια από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί. Υπάρχουν διάφορες δοξασίες και προκαταλήψεις ε, ιονή, ε, γρουσουζιά και άλλα πράγματα που επικρατούν στις κοινωνίες αυτές και θεωρούνται ως εκ τούτου ε, επικίνδυνα αυτά τα δύστιχα άτομα που πάσχουν από αλφισμό θεωρούνται πολύ επικίνδυνα και ως εκ τούτου η κατάσταση γίνεται πολύ επικίνδυνη για αυτούς ε, οι δυνατότητες είτε για την ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την ε, διατήρηση, την βελτίωση ενός κοινωνικού επίπεδου είναι μηδαμινές. Υπάρχει αδύρυτη ανάγκη για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και βεβαίως οι προσπάθειες από τις αρχές της ποινική δικαιοσύνης για διώξεις εις βάρος εκείνων που έχουν διαπράξει βίες πράξεις βάρος ατόμων μαλφισμού έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα εκ μέρους της ομάδας συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερος, καθώς μάλιστα είμαι και ο ίδιος γιατρός, ε, που μπορούμε να ε, φέρουμε το ψήφισμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το εγκρίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Χόιμπουχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η βία εις βάρος των ανθρώπων με αλφισμό είναι αδιανόητο, ε, ε, αδιανόητη. Έχουν προβλήματα στο σχηματισμό της μελατονίνης και αυτό οδηγεί και μέχρι στον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και σε τελείως πρακτικά προβλήματα, γιατί δεν τους επιτρέπεται η ομαλή πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική θρησκευτική περίθαλψη όπως μόλις τώρα αναφέρθηκε ή η πρόσβαση σε απλά ε, προϊόντα όπως το αντιλιακό. Πολύ συχνά ε, κινδυνεύουν ε, και νοσούν από από δερματικές παθήσεις και κυρίως καρκίνο του δέρματος. 9 από 19 άτομα με ε, αλφισμό στην Τανζανία δεν φτάνουν στην ηλικία των 30. Πολλές φορές πέφτουν θύματα βίων επιθέσεων. Ε, τα θεωρείται από τις δοξασίες της ε, Αφρικής ότι τα, ένα κομμάτι από το σώμα τους μπορεί να έχει μαγικές ιδιότητες και πολλές φορές τους κατακρεουργούν τα παιδιά δεν έχουν δυνατότητα στην, πρόσβαση στην εκπαίδευση, κινδυνεύουν όλα τα άτομα με αλφισμό και ιδιαίτερα στο Μαλάουι όπως έχουμε δει και τα θύματα, χρειάζονται καλύτερη προστασία Ιδιαίτερα θέλω να χαιρετήσω το ότι έχουν γίνει εξαγγελίες μέτρων στο Μαλάουι και την Τανζανία εκ μέρους των κυβερνήσεων αλλά και από τα Ηνωμένα Έθνη έχουμε ακούσει εξαγγελίες, έχουμε ακούσει για ε, περιφερειακές πρωτοβουλίες και Βεβαίω περιμένουμε μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξει τις ε, προσπάθειες για την εξασφάλιση φερρυπίν ε, κατάρτιση για τους αστυνομικούς άντρε και γυναίκες την ενίσχυσή του εκεί. Το Κοινοβούλιο δίνει την ε, δίνει, δίνει φωνή στους ανθρώπους αυτούς σήμερα. Ελπίζω στο μέλλον να μην χρειαστεί να συζητήσουμε άλλο ψήφισμα για τα προβλήματα των ανθρώπων με αλφισμό. Πιστεύω να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με το καλό αυτό ψήφισμα τους ανθρώπους στην Αφρική. Ευχαριστώ πολύ. Κορά, Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την είπα το εκπρόσωπο. Όταν μιλάμε για τους Αλμπίνους στο Μαλάουι, και στην περιοχή αυτή ευρύτερα έχει δημιουργηθεί μια απαράδεκτη, παράλογη κατάσταση, υφίστανται ακροτηριασμούς, βασανιστήρια, ακόμα και μεταθάνατον, θάνατον, όπως είπε η συνάδελφος, ε, τα οστά τους πολλούνται διότι υποτίθεται μπορεί να χρησιμεύσουν ως ανφυλακτά και Επίσης πιστεύετε ότι πρέπει να βιάζονται οι γυναίκες αλμπίνο διότι έτσι θα αποκτήσουν ανοσία για το AIDS αυτοί που το κάνουν. Νομίζω ότι εμείς έχουμε σχέσεις διεθνούς συνεργασίας με το Μαλάουι και μέσω της Συμφωνίας του Κοτονού και θα πρέπει εμείς να προστατεύσουμε αυτή την μειονότητα η οποία γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ουσιαστικά από εγκληματικές συμμορίες που ωφελούνται από αυτούς και οικονομικά. Σας ευχαριστώ. Κύριος Φίσας, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτό που συζητάμε σήμερα πρέπει να βοηθήσει για να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα στι αφρικανικέ χώρε εκεί όπου παρουβιάζονται τα δικαιώματα των ε, αλμπίνος τα οποία υποφέρουν από τι χειρότερε διώξει και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Ε, λεκτική βία, αλλά όχι μόνο και φυσική βία μέχρι και δολοφονίε. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και συμβαίνουν όχι μόνο στο Μαλάου, αλλά και στην Τανζανία, το Μουρούντι, στη Μοζαμβίκη και στην Κένια. Τα άτομα Αλμπίνο. Ε, υποφέρουν από διακρίσεις κοινωνικές αλλά και όχι μόνο και στην περίθαλψη. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ε, καρκίνου του δέρματος, όμως πολύ δύσκολα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία, οπότε είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για να σταματήσει αυτή η τραγική κατάσταση, αλλά δεν φτάνουν. Πρέπει να ληφθούν μέτρα πρόληψης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και να διώκονται οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων. Τα άτομα αυτά είναι πολύ ευάλωτα, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, πρέπει να τα στηρίξουμε για να μπορέσουν να διώξουν με τη σειρά τους ε, τους εγκληματίες. Ευχαριστώ κύριε Σπαντσέλη, έχει το λόγο. Η σιωπηλή τραγουδία των Αλμπίνων στην Αφρική παίρνει πάρα πολλές μορφές και σε επίπεδο σωματικό με άσκηση βίας βάρος τους, με ακροτηριασμούς λόγω πραγματικά ε, απαράδεκτων προκαταλήψεων που αναγνωρίζουν υποτίθεται ε, πάρα πολύ ε, φανταστικές ικανότητες ή προβλήματα στους ανθρώπους αυτούς και αυτό οδηγεί φυσικά και στην προσπάθεια αποκλεισμού τους από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τον αποκλεισμό τους από τον χώρο της εργασίας, Πρέπει να σταματήσουν αυτά τα απαράδεκτα εγκλήματα εις βάρος των Αλμπίνο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις αυτές και να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο από την κοινωνία. Πρέπει να πιέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο σας. Πρόεδρε, όταν γεννιέται ένα παιδί παντού, όταν γεννιέται ένα παιδί παντού οι γονείς του χαίρονται. Αλλά όχι στο Μαλάουι αν γεννηθεί λευκό παιδί. Γιατί τότε αισθάνονται ότι τους έχει τιμωρήσει ο Θεός. Τα παιδιά αυτά τα βλέπουν με πολύ μεγάλη καχυποψία. Πρόκειται για δοξασίες συνδυασμένες ε, με τα ε, διδάγματα των ε, μάγων γιατρών που λένε στον κόσμο ότι έχουν μαγικά, μαγικές ιδιότητες η τα κομμάτια του σώματος των ατόμων με αλφισμό. Μέχρι και για 75.000 δολάρια το κόκαλο, το οστό είναι η τιμή της αγοράς. Το φαντάζεστε αυτό. τα κορίτσια, οι γυναίκες με αλφισμό πέφτουν θύματα βιασμού γιατί οι άντρες ε, πιστεύουν ότι τους προσφέρουν έτσι ε, αγωγή κατά του έτσι προστασία κατά του έτσι Αυτό είναι απαραίτητο να πέφτουν θύματα δίωξη, βίας, ε, κυνηγιού ακόμη αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Σάντσε Κάλντεντε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Αλμπίνος στην Αφρική αντιμετωπίζουν ακραία δίωξη και παραβίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Υπάρχει διάκριση στην κοινωνία γενικευμένη, αλλά είναι και θύματα δολοφονιών και ακροτηριασμών. Οι απειλέ αυτέ οφείλονται σε προκαταλήψει, ότι έχουν μαγικέ ιδιότητε τα άτομα αυτά. Πιστεύουν ότι αν υπάρχουν σεξουαλικέ σχέσει με αυτού μπορούν να θεραπευτούν από το AIDS. Οπότε πολλοί τους δολοφονούν για να πάρουν κομμάτια από το σώμα τους γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα έχουν πλούτο και υγεία. Εμείς στην εξωτερική μας δράση μερικές φορές επιδεινώνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, τις κοινοφελείς υπηρεσίες, στις χώρες του Νότου με εμπορικές μας πολιτικές που είναι άδικες απέναντί τους. Ο πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα είναι να ενισχύσουμε τι κοινοφιλεί υπηρεσίε στι χώρε αυτέ, την εκπαίδευση, για να σταματήσουν αυτοί οι μύθοι χρειάζεται εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινοφελείς υπηρεσίες ποιότητας. Αυτό χρειάζονται αυτές οι χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ομιλητέ εκ μέρου των ομάδων Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κύριο Πρέντα έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου στην συζήτησή μας και να προσθέσω στη συνέχεια ότι ζήτησα από την ομάδα μου να προωθήσουμε ένα ψήφισμα κατεπήγων για την κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική. Με χαρά λοιπόν διαπιστώνω την υποστήριξη που προσφέρεται από τους λοιπούς συναδέλφους. Πρέπει να πω ότι ένα έναυσμα για την πρόταση αυτή ήταν η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που κατατέθηκε πριν από, πριν από λίγο καιρό, ιδίω για το Μαλάουι, αλλά όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, βίες επιθέσεις, αποτρόπαιοι φόρνοι αφορούν και άλλες χώρες, Τανζανία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού. Σε όλες αυτές τις χώρες σημειώνονται φρικτά εγκλήματα κατά των ε, ανθρώπων που πάσουν από αλφισμό. Και αυτή ήταν η ιδέα και το έναυσμα για την συμπερίληψη της συζήτησης στην ημερήσια μας διάταξη. Σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν για τη συμμετοχή των συναδέλφων και την ευαισθησία που δείχνουν και την ανησυχία για τα άτομα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, και τώρα η κυρία Κέντζη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το να γεννηθεί κανείς αλμπίνο σε ορισμένες χώρες της Αφρικής σημαίνει ότι κινδυνεύει να πεθάνει, κινδυνεύει να ακροτηριαστεί σε καθημερινή βάση. Το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτόν τον αποχρωματισμό και υφίστανται δυστυχώς ε, κάποιες φρικτές πρακτικές στιγματίζονται σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση όχι μόνο του Μαλάουι αλλά και όλων των χωρών όπου διαιωνίζονται αυτές ε, οι πρακτικές να υπάρξει μια πολιτική καταπολέμησης του αποκλεισμού, μια στρατηγική αποκλεισμού των διακρίσεων ουσιαστικά όλοι θα πρέπει να κρίνονται με ισότιμο τρόπο, όλοι θα πρέπει να γίνονται, να υπάρχει σεβασμός χωρίς διακρίσεις εις βάρος τους. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Τζέμς. δύο λεπτά. Τις τελευταίες εβδομάδες στο Βρετανικό τύπο είδαμε πολλές ε, περιπτώσεις όπου οι δοξασίες ε, και τα ε, μαγικά, μαγικές μέθοδοι είχαν συνέπειες για τη ζωή των ατόμων με αλφισμό όπως βέβαια και γενικότερα ζητήματα απασχόλησης εκπαίδευσης και ε, ευημερίας πλήττονται λόγω ακριβώς αυτής της αποτρόπαιης συμπεριφορά απέναντι στου άτομα με αλφισμό. Πρέπει ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει πάνω από όλα το πρόβλημα των αποτρόπαιων οικονομικών φραγμών ει βάρο των κρατών τη Αφρική. Μόνο αυτά που θα επιτρέψουν δηλαδή, την οικονομική και κοινωνική ευημερία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, θα δώσουν ένα τέρμα στι δοξασίε, τι προκαταλήψει και τι μαγικέ μεθόδου και έτσι θα δώσουν μια ευκαιρία σε όλου του πολίτε των Αφρικανικών κρατών και όχι μόνο στα άτομα με αλφισμό. Η Βρετανική κοινοπολιτεία από εδώ και μπρο θα δράξει τα ενία για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, αλλά καλό και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κοιτάξει τι είδου πρακτικέ έχει αναπτύξει με την Αφρική, γιατί δεν βοηθάει καθόλου την κατάσταση των ατόμων με αλφισμό, την κατάσταση των ατόμων με φτώχεια, την κατάσταση γενικά των Αφρικανών. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Κόρμιν και ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, φοβάμαι ότι νιώθω κάποια αηδία με αυτή τη συνένεση που δημιουργείται. Νομίζω όλα αυτά είναι βλακίες, όλα αυτά είναι ανοησίες. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Οι Αμερικανοί έχουν προβλήματα στην Αφρική αγόρασαν ένα κομμάτι γης και δημιούργησαν τη Λιβερία. Ίσως πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο, να δημιουργήσουμε ένα κράτος όπου μπορούν να ζουν οι αλφικοί. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι θετικό για την κατάστασή τους. Αυτά τα οποία λέμε τώρα δεν οδηγούν σε τίποτα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως είναι για τα μπάζα. Πρέπει να καταστραφεί. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Ο κύριο Βέντα ακολουθεί από την ομάδα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπος, ο αλφισμός για λόγους οι οποίοι είναι άγνωστοι αποτελεί ένα πρόβλημα στην ε, Μεσημβρινή Αφρική, ίσως γιατί είναι πιο διαδεδομένο αυτό το πρόβλημα από ό,τι σε άλλες χώρες του κόσμου. Οι αλφικοί ζουν σε συνεχή φόβο γιατί κινδυνεύουν να κακοποιηθούν. Τα παιδιά μπαίνουν σε ειδικά ιδρύματα για να προστατευτούν. Αλλά πάντα υπάρχει και επικρέμαται η απειλή εναντίον της ζωής τους όσο μεγαλώνουν. Το Μαλάου είχε μια μεγάλη έξαρση επιθέσεων κατά των αλφικών. Αυτό καταδεικνύει ότι έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα και ένα μεγάλο κίνδυνο για αυτό το τμήμα των πολιτών του Μαλάου. Πρέπει οι τοπικές αρχές να κάνουν όλα τα απαραίτητα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το δικαίω, τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων εκεί και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και άλλες χώρες να παρακολουθήσουν αυτά τα οποία συμβαίνουν σε χώρες όπως το Μαλάου στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τα αφρικανικά κράτη για να σταματήσει αυτό το βαρβαρικό έθιμο. Κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε οι Αλμπίνο στο Μαλάουι δολοφονούνται, ακροτηριάζονται και τα οστά τους πολλούνται. και η Amnesty International επίσης καταγγέλει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση όπου τμήματα του σώματός τους χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ε, λαϊκών φαρμάκων και ουσιών, εν πάση περιπτώσει, ε, που υπόκεινται σε απαράδεκτες προκαταλήψεις. Υπάρχουν απαγωγές, υπάρχουν συνεχείς δολοφονίες και ζούνε ε, στα πλαίσια ε, του τρόμου σε καθημερινή βάση. Πρέπει λοιπόν να αναλυφθεί η δράση έτσι ώστε να υποχρεωθεί η δημοκρατία του Μαλάουι να προστατεύσει τους Αλμπίνο και να προστατεύσει και το δικαίωμά τους στη ζωή. Ευχαριστώ. Και έχουμε φτάσει στο τέλος του καταλόγου με τον κύριο Επιτήριο από τους μη με Ένα λεπτό. Οι οποίε ε, συμβαίνουν ορισμένε από τι πιο ακραίε μορφέ ρατσισμού και παραβιάσεω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια τέτοια περίπτωση είναι οι διωγμοί που υφίστανται τα άτομα με αλθισμό σε διάφορε αφρικανικέ χώρε και κυρίω στο Μαλάουι. Όπω γνωρίζετε πολύ καλά, οι δυστυχεί αυτοί οι άνθρωποι κακοποιούνται, γίνονται ε, θύματα επιθέσεων υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό υφίστανται ακροτηριασμούς βιασμούς γίνονται θύματα προκαταλήψεων και δολοφονούνται. επειδή είμαι αντίθετο σε κάθε διάκριση η οποία βασίζεται στην φυλή το φύλο το χρώμα και τις ιδιαιτερότητες καταδικάζω απερίφραστα αυτή τη ρατσιστική συμπεριφορά των αφρικανικών κυβερνήσεων και κυρίως της του μαλάουι απέναντι στα άτομα με αλφισμό. δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό κυβερνήσεις αφρικανικές οι οποίες διαμαρτύρονται για τον ρατσισμό εις βάρος των αφρικανών να συμπεριφέρονται με τρόπο που αρνούνται στους άλλους να συμπεριφέρονται. επιπλέον εκφράζω την ε, ανησυχία μου μήπως μέσα στις εκατοντάδες χιλιάδες παρανόμων μεταναστών που έχουν κατακτήσει την ελλάδα και την ιταλία υπάρχουν άνθρωποι με τέτοιες ακραίες και επικίνδυνες τάσεις. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Περνάμε τώρα στην διαδικασία Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο σε όλους που το έχουν ζητήσει. Το λόγο ο κύριος Κέλλης πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήταν κάπω παράξενα αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον κύριο Κόρβιν Μίκε. Είπε ότι θα πρέπει να καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλλά από την άλλη πλευρά η Ένωση που θέλει να καταστρέψει θα πρέπει να αγοράσει ένα κομμάτι γης για να εγκαταστήσει εκεί τους αλφίκους. Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Όταν δείτε το πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό βασίζεται αποκλειστικά στη δυσυδαιμονία. Αντί λοιπόν να κάνουμε κάτι άλλο, θα πρέπει να ξεπεράσουμε τη δυσυδαιμονία. Ίσως με τα Ηνωμένα Έθνη θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ε, στο Μαλάουι και σε άλλες χώρες συνδιασκέψεις και παιδεία για να καταλάβουν όλοι ότι αυτές οι δυσδαιμονίες δεν έχουν καμία βάση και ότι η Αλφική είναι ίδια με όλους τους άλλους ανθρώπους. Αν λοιπόν αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, έτσι νομίζω μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που τυπώσατε μια διαφορετική άποψη. Ο Μαριάς τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε στηρίζω το κοινό ψήφισμα το οποίο έχω συνυπογράψει και εγώ. οι διακρίση σε βάρος των ατόμων που πάσχουν από λευκοπάθεια και η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους αποτελούν συχνό φαινόμενο σε πολλές χώρες της αφρικής και κυρίως στο μαλάουι το οποίο είναι μια από τις φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρε παγκοσμίω, με το 50,7% του πληθυσμού να ζει κάτω από τα όρια τη φτώχειας σύμφωνα με την αστυνομία του μαλάουι το 2014 καταγράφηκαν τουλάχιστον 65 περιστατικά βίας κατά ατόμων που πάσχουν από λευκοπάθεια εκ των οποίων 18 άνθρωποι δολοφονήθηκαν ενώ τα περιστατικά παράνομου εμπορίου οστών και μελών του σώματος των ατόμων αυτών είναι πολύ συχνά απέναντι στη διαρκώ αυξανόμενη καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μαλάουι η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να προστατεύσει του ανθρώπου που πάσχουν από λευκοπάθεια και να καταδικάσει τι δολοφονίε και την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων. επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίξει την ίση πρόσβαση αυτών των ατόμων σε υγειονομική περίθαλψη εκπαίδευση καθώ και σε κοινωνική και νομική προστασία. ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Μογκαντίνη έχει το λόγο. Κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ νιώθω την ίδια έκπληξη, όπως την εξέφρασε και η συνάδελφός μας, Κάθε φορά που κάποιο λέει τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, δεν μπορούμε συγχρόνω να λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Ήδη είναι αντιφατικό κάποιο ο οποίο δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται σε αυτό το ημικύκλιο. Ούτω ή άλλω. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την ε, ομόφωνη θέση σας για αυτό το σημαντικό θέμα. Τα δύο τελευταία χρόνια το Μαλάο έχει αντιμετωπίσει μια σημαντική αύξηση σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον ε, πολλών αλφικών, κυρίως παιδιών βίες επιθέσεις και εγκλήματα, απαγωγές, δολοφονίες. Όλη αυτή η βία καταδεικνύει ότι υπάρχουν υποβόσκοντα σοβαρά προβλήματα ε, διακρίσεων αντίον αλφικών σε πολλά μέρη της υποσαχάριας Αφρικής, όχι μονάχα στο Μαλάουι αλλά και στη Μοζαβίκη, το Μπουρούντι και άλλες χώρες. Εμείς έχουμε στις 11 Ιουνίου την Διεθνή ημέρα ε, συνειδητοποίησης για τους ε, αλφικούς. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα για να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες μας τα προβλήματα αυτά και επίσης διορίστηκαν οι πρώτοι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της αντιμετώπισης των προβλημάτων των Αλμπίνων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε αυτή την κοινότητα και εγώ προσβλέπω στο να συνεργαστώ μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτό το εγχείρημα το οποίο είναι εγχείρημα συνειδητοποίηση αλλά και παιδεία, όχι μόνο για το Μαλάουι αλλά και σε άλλε χώρε. Πρέπει λοιπόν με τι δεσμεύσει αυτέ να κάνουμε όλα τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε του αρθικούς οι οποίοι βρίσκονται σε σε κίνδυνο. Θα πρέπει να σταματήσει η διάκριση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές δυνητική διάκριση. Ζητούμε λοιπόν από τι κυβερνήσει των χωρών αυτών που γίνονται τέτοιε επιθέσει να οδηγήσουν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τα προβλήματα αυτά και να γίνουν κατανοητά όλα αυτά ακόμα και σε επίπεδο οικογένεια, ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει σεβασμό τη ταυτότητα και τη αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών. Θα πρέπει να σταματήσουν λοιπόν και οι διακριτικέ μεταχειρήσει εναντίον των ανθρώπων αυτών, ώστε να έχουν την κατάλληλη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την παιδεία <clears throat> και την απασχόληση. Αυτό δεν είναι ένα θέμα μοναχα του Μαλάουι, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά πολλές περιοχές της Αφρικής, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μεταλαμπάδευση βελτίστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της Αφρικής για την προστασία των δικαιωμάτων των αλφικών και την ε, αποτροπή διαμεθοριακών διώξεων και εγκλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των αντιπροσωπιών μας θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τις τοπικές κυβερνήσεις και με τις κοινωνίες των πολιτών των χωρών αυτών. Πιστεύουν ορισμένοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε τι κοινωνικέ πρακτικέ στι χώρε αυτέ, τι δυσαιμονίε, την καχύποπτη στάση εναντίον των αρφικών. Εγώ διαφωνώ. Νομίζω ότι αν έχουμε μια συνεργατική και κοινή προσέγγιση μαζί με του εταίρου μα, μπορούμε να αλλάξουμε και τι νοοτροπίε. Πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειές μα να αλλάξουμε σε επίπεδο καθημερινότητα τις ρίζες αυτής της ε, αποτρόπιας συμπεριφοράς η οποία πρέπει και να αλλάξει το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τα καθησυχαστικά σας λόγια. Θέλω να πληροφορήσω το κοινοβουλίο μας ότι έχουμε λάβει 7 ψηφίσματα για την λήξη της συζήτησης